εκπέμπουμε αυτό το αίτημα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η συνάδελφος ε, κυρία Λάρα Κόμη μου υπέβαλε ένα αίτημα υπεράσπισης της ε, κοινοβουλευτικής της ασυλίας ε, και ο κ. Γκαμπριέλη Αλμπερτίνη. Σύμφωνα με το άρθρο 6, πράγραφος 3 του κανονισμού, έχουν σταλεί αυτές οι αιτήσει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και από την ομάδα των Πρασίνων